Συνάδελφοι, συνεχίζουμε μετά την συνάντηση και κλεισμένων των θυρών. Ήταν μια καλή ευκαιρία για να δούμε ακριβώς ποια είναι η πρόοδος που έχει συντελεστεί σε σχέση με την κτηριακή πολιτική. Λοιπόν, ε, θα ακούσουμε την ανακοίνωση των διευμηνέων για μια ακόμη φορά, λέει ευγενικά ο πρόεδρος, τον ευχαριστούμε. Είναι η τρίτη βδομάδα όπου συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας ε, απέναντι στα νέα μέτρα τα οποία εφαρμόζει η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία επαφή με τον Γενικό Γραμματέα. Δυστυχώς ε, οι, επι, επιστρατεύσεις συνεχίζονται για πολλούς από τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να είστε σύντομοι γιατί 12.30 θα σταματήσουμε τις εργασίες μας. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, λέει ο Πρόεδρος, δεκτή ημερήσια διάταξη. Η συνάντηση των συντονιστών της 16ης Μαΐου περιλαμβάνεται στα πρακτικά και οι αποφάσεις τους θεωρούνται δεκτές αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Σχετικά με τα πρακτικά της 22ης ε, ε, Δευτέρας συγγνώμη, Μαρτίου και του Απριλίου, ε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, γίνονται δεκτές. Θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες για την κτηριακή πολιτική καταρχάς η ψηφοφορία αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα για την συνάντηση της 28ης Ιουνίου. Γι' αυτό θα περάσουμε τώρα στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαρίθμου 2 Μουρεσάν Εφόσον έχετε τις κάρτες σας, παρακαλώ να είστε έτοιμοι. Θα γίνει μια δοκιμαστική ψήφος, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Sur le rapport De budget modificatif numéro... Τώρα λοιπόν για, το, για την διορθωτική επιστολή 2, τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Με μια προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, δεκτό για το σύνολο του κειμένου, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίας 30 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή συγχαρητήρια στον Γενικό Εισηγητή, τον κύριο Μουρεσάν. Τώρα περνάμε στην επόμενη έκθεση για τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα συστήματα πληροφορικά για τα σύνορα και τη χορήγηση θεωρήσεων. Είναι τα σημεία 8 και 9 δύο προτάσεις του κυρίου Κέλμελ. Διαλειτουργικότητα λοιπόν συστημάτων, συνεργασία αστυνομική, συνεργασία δικαστική και επίσης ε, διαλειτουργικότητα των συστημάτων χορήγησης θεωρήσεων. Θα δώσω το λόγο σύντομα όμως στον εισηγητή μας, τον κύριο Κόλμελ, ο οποίος θα μας διαφωτίσει για τις τροποποιήσεις τις οποίες έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας κάνει παρατηρήσεις για τις ψηφοφορίες σήμερα, αν πιστεύετε ότι μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα. Έχετε το λόγο κύριε Κόλμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να καταχαστώ του διαθεσίμου χρόνου. Νομίζω ότι έχουμε ε, κάνει επανειλημμένες συζητήσεις, έχουμε εμβαθύνει στις εκθέσεις αυτές. Είναι εκθέσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την ε, ασφάλεια, αλλά είναι επίσης ε, κάτι το οποίο κοστίζει. Πρέπει να επενδύσουμε μισό εκατομμύριο Νομίζω όμως ότι τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν σωστά και δικαιολογημένα. Να θυμίσω ότι χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέους αριθμούς Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της, δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο ε, δυστυχώς βέβαια στο παρελθόν οι πολλές αλλαγές οδηγούσαν σε πολύ πιο ακριβές προτάσεις. Οι υπολογισμοί που γίνονται ε, για τη χορήγηση θεωρήσεων απαιτούν 33,6 εκατομμύρια επιπλέον για την αγορά λογισμικών ε, και συνολικά θα χρειαστούν θα χρειαστεί ένα ποσό ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι κρίσιμο στην παρούσα φάση είναι να ελέγχουμε από πάρα πολύ κοντά αυτούς, αυτούς, αυτές τις προμήθειες και τις διαδικασίες προμηθειών έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να καταλήγουμε στις πιο οικονομικές λύσεις έτσι ώστε στην τελευταία στιγμή να μην ε, υπάρχουν ανατιμήσεις και αυξήσεις των απαιτούμενων ποσών. Merci, Monsieur Colmel. Donc, nous pouvons passer au vote. Ευχαριστώ κύριε Κόλμελ. Τροπολογία 8. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. 9 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Το 10 έχει αποσυρθεί. 3 υπέρ. Έχει καταπέσει το 3. Όχι, πρέπει να ψηφιστεί. Το 3 λοιπόν ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 11 έχει αποσυρθεί. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Το σύνολο του τοπολογημένου κειμένου τώρα με ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρα τις ψηφοφορίες, 30 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή, συγχαρητήρια στον κύριο Κόλμελ. Για το δεύτερο κείμενο, διαλειτουργικότητα του συστήματος ενημέρωσης συνοριακών ελέγχων και χορήγησης θεωρήσεων. Τροπολογία 8. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 10 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έντεκα. αποσύρεται. Πέντε. υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 23-12. Τροπολογία υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. 30 υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Νιριάντα. για την αύξηση της χρηματοδότησης ε, και για την υποστήριξη των ε, διαρθρωτικών αλλαγών. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-14. Λοιπόν, τότε πρέπει να ψηφίσουμε μία-μία τις τροπολογίες του συμβιβαστική. Τροπολογία 11. Προφορική τροπολογία αφορά για τη σύγκληση in και out. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. πέρας, Απορρίπτεται. 22 ψήφι κατά, 14 υπέρ. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος της τροπολογίας 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 21, 21 ψήφοι κατά, 14 υπέρ. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-14. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική, συγγνώμη, τροπολογία 19, ο διορθώνει ο πρόεδρος, συμβιβαστική 2, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε μία-μία τις τροπολογίες που κάλυπτε αυτός ο συμβιβασμός, δύο. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρι... ε, απορρίπτεται, συγγνώμη, 17, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, Τροπολογία... ε, συγγνώμη, τμήμα 2, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. υπαριθμών 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρα... Μία-μία τις τροπολογίες. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επτά με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Απο, αποχές απορρίπτεται. Για το 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε μία-μία τις τροπολογίες που κάλυπτε, τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Καταπίπτη. Πάμε στην 29 υπέρ. Καταπίπτει και αυτή η τροπολογία και η 30 καταπίπτει. Άρα Πάμε στην 9. Και αυτή καταπίπτει. Πάμε στη 10 άρα. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Νηριάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης, ε, την ε, έκθεση ε, του κυρίου Λαμασού για την Ερφρός, τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Το 7 και το 8 και 8 καταπίπτουν. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 έχει αποσυρθεί και 11. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Έχει αποσυρθεί. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 15 υπέρ. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας.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 Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σύνολο του κειμένου τώρα με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται 31, 3 και 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Λαμασού. Nous avons maintenant à nous prononcer sur... Euh, Πάμε τώρα σε δύο αιτήσει μεταφοράς. Ο Μούρισαν είναι εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλημερίζω συνάδελφοι. Απόφαση 10 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια μεταφορά συνέπεια της ψηφοφορίας της έκθεσης Λαμασού. 9,89 εκατομμύρια για απολυθέντες εργαζομένους από εταιρείες όπως η ΕΦΡΑΣ και η Γαλλική ΔΕΗ. Ελπίζω να υπερψηφίσετε την πρόταση. Θα ψηφίσουμε λέει ο Πρόεδρος για την συγκεκριμένη πρόταση του κυρίου Μουρεσάν 10 του 18. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 23 υπέρ, 3 κατά. Δεύτερη μεταφορά, ο Γενικός Εισηγητής. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, Πρόεδρε. Διοικητικές δαπάνες. Απλό θέμα. 14,1 εκατομμύρια μεταφορές ανάμεσα στους διαφορετικές γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν δύο πηγές για τα χρήματα αυτά. Πρώτα ποσά τα οποία δεν είχαν κατανεμηθεί για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες και δεύτερον αναθεώρες ανάγκες και αναδιοργανώσεις στο DG Level για αποστολές και πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά. Πηγαίνουν στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και στην ε, Γενική Γραμματεία για Συστήματα Πληροφορικής. Στην DG Home επίσης για θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, DigiNear για την Ανατολική και Νότια Γειτονία, DigiMove Move, αποστολές στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της Συμφωνίας Open Skies, DGCOM για αποστολές. Λοιπόν, έχοντας εξετάσει ακριβώς την προέλευση και την κατάληξη των προορισμό των ποσών αυτών, ζητώ να γίνει δεκτή η πρόταση για τη μεταφορά 14,1 εκατομμυρίων. Θέτω σε ψηφοφορία την πρόταση, λέγει ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρόεδρο, οι διευμηνήσεις ζητούν να πατήσετε το κουμπί του μικροφόνου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είχε αρχίσει η ψηφοφορία. Ζητώ ε, σε αυτούς που δεν με άκουσαν να ψηφίσουν. Πέρα της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 3 κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Μουρεσάν. Ashworth. Θέλετε να μας παρουσιάσετε τις δικές σας συστάσεις για την μεταφορά ε, της ε, Επιτροπής Περιφερειών όπως επίσης και του ελεγκτή προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού και σχετικά και με το ε, οργανόγραμμα. Έχετε το λόγο. Δύο θέματα καταρχάς για τον ελεγκτή προσωπικών δεδομένων 700.000 ευρώ από τις αμοιβέ ε, στις ε, συμβάσεις προσωπικού. 15 επιπλέον συμβόλαια για το νέο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και κάλυψη εξόδων που δημιουργούνται από άδειε κοίησης. Νομίζω ότι είναι μια λογική πρόταση και νομίζω ότι η μακροπρόθεσμα εξοικονομεί χρήματα. Δεύτερο αίτημα, πάντα από τον ελεγκτή προσωπικών δεδομένων. Μία μεταφορά θέσης AST1 σε AST2. Και εδώ συστήνω την έγκριση δεν έχω τεχνικές ε, γνώσεις ειδικά γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε μπορείτε να συνδέσετε και τα δύο αιτήματα μεταξύ τους και να κάνετε μία ψηφοφορία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τελευταίο σημείο. Έτοιμα της Επιτροπής Περιφερειών θέλουν να κάνουν μια μεταφορά. Ζητήσαμε περισσότερες πληροφορίες από αυτούς. Περιμένουμε τις πληροφορίες αυτές. Σας προτείνω λοιπόν να γίνει η ψηφοφορία αυτή στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η τρίτη μεταφορά αναβάλλεται στην επόμενη συνάντηση και για τις δύο πρώτες μεταφορές, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, γίνονται δεκτές θα δώσω τώρα το λόγο στη Μόνικα Χολμάγερ για την κτηριακή πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σύντομη εισαγωγική ενημέρωση. Η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιούλιο για αυτό το θέμα. Πρόκειται για το κτίριο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής EBA στο Παρίσι. Στις 9 Ιουλίου που θα κληθούμε να ψηφίσουμε θα παρακαλέσω να μας ενημερώσει η Τραπεζική Αρχή για το τι συμβαίνει με την υποστήριξη της Βρετανικής κυβέρνησης ε, για τη μελλοντική μοίρα του τωρινού κτηρίου. Πώς το βλέπει εκεί, ε, γιατί το κόστος που έχει προκύψει μέχρι ετησίως είναι 3,7 εκατομμύρια για το συγκεκριμένο κτίριο στη Βρετανία και σε μια δεκαετή περίοδο μέχρι το 2026 θα πρέπει να πληρώνουμε ε, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ε, κάποιος νέος ε, νοικιαστής. Η μελλοντική κατάσταση πώς διαγράφεται λοιπόν. Ο οργανισμός EBA προκήρυξε και πάλι διαγωνισμό παρόλο που είχε προκήρυξει η γαλλική κυβέρνηση προηγουμένως και είχε βρεθεί και κτίριο το οποίο ήταν και φθηνότερο και καταλληλότερο και το είχε αξιολογήσει θετικά και η γαλλική κυβέρνηση. Η μετακόμιση θα γίνει ε, στο, ε, στην περιοχή Defense, ε, στον 24ο με 27ο όροφο του ενός πύργου, 9 ετής μίσθωση 6 ε, συν 3 ε, η τραπεζική αρχή ε, διδάχτηκε από την περίπτωση του Λονδίνου ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί για διάφορες αντικσότητες και αν αλλάξει τίποτα στο καθεστώ θα πρέπει να μπορεί να αποσυνδεθεί από τη σύμβαση. 560 τετραγωνικά περίπου είναι, έχουν ε, και τους υπαλλήλου που θα πρέπει να μετακομίσουν εκεί ε, και ε, θα μεταξελιχθεί και το όργανο αυτό. 1,952 εκατομμύρια είναι το μίσθωμα ετησί και 22 μήνες δεν μπορεί να νοικιαστεί αυτό το κτίριο. 1,5 ε, εκατομμύριο θα δώσει η γαλλική κυβέρνηση για τα αρχικά έξοδα και 7 εκατομμύρια επιδότηση ενοικίου. Ε, σύνολο το κόστος για 34 μήνες, δηλαδή μια έκπτωση ενοικίου 350.000 ευρώ το μήνα οικονομική υποστήριξη από τη γαλλική κυβέρνηση υπάρχει. Αυτή είναι εξάρτητη από το κτίριο που επελέγει. Την άλλη εβδομάδα ε, θα ελεγχθεί ο φάκελος, ε, θα το κάνω σε συνεργασία με το Σκιώδης, θα μελετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ενδιαφέρεται πολύ να μας ενημερώνει εγκαίρως και εκτενώς και έχω την αίσθηση ότι σε αντίθεση με την περασμένη κατάσταση στο Λονδίνο που ήταν όλα καινούρια ε, για τους υπαλλήλους, τώρα είναι πιο διαρθρωμένη και πιο μεθοδική και συστηματική η προσέγγιση. Οπότε όλα αυτά ε, διαγράφονται πάρα πολύ και διαφαίνονται πάρα πολύ θετικά. 9 ή 10 Ιουλίου θα ψηφίσουμε. Και όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες είμαι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ευχαριστώ τη Μονίκα Χολμάιερ για την ανακοίνωση αυτή. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Θα το συζητήσουμε και από την άλλη εβδομάδα μετά. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς το λόγο γι' αυτό. Όχι. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Που είναι και επίκαιρο γεωπολιτικά. Η πολιτική προπολογισμό θέλησε να ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το θέμα της απόφασης ε, κατοξιδότησης 6 Ιουνίου που προσθέτει το Ιράν ε, στις χώρες που ενισχύει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, ο κύριος Φλέκενστάιν είναι μόνιμος εισηγητής για το Ιράν και μέλος της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Ε, έχει προσκληθεί εδώ και άλλα μέλη της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Ο κύριος Λεβαντόφσκι είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου με το Ιράν και θα μπορέσει να μας διαφωτίσει σχετικά. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους ομιλητές για τρία λεπτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την κυρία Άννα η οποία είναι αρμόδια για ε, την μονάδα, το τμήμα ΕΚΦΙΝ L1, L1 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανάπτυξη. Ο κύριος Μπερτράν Τεβασιέρ, Γενικός Διευθυντής της Αρμόδιας Οικονομικής Διεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε τον κύριο Τρότσεν Μπάρκρεφτ και συγγνώμη αν κατακρεούρισα το όνομά σας είστε αρμόδιος για την Task Force Iran και στη διάθεσή μας για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Η κυρία Άννα Κρυζανόφσκα έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια για την εξουσιοδότηση πράξη, της οποίας ε, ο σκοπός είναι από τον κατάλογο των ενδεχομένως ε, επιλέξιμων χωρών ε, για την χορήγηση εγγύησης στις πλήρως επιλέξιμες χώρες, στην κατάσταση των πλήρως επιλέξιμων χωρών. Στις 6 Ιουνίου εγκρίθηκε αυτή η πράξη. Η διαδικασία προβλέπεται στην απόφαση ΕΛΕ ε, στις 14 Μαρτίου ε, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα ήθελα να αναφερθώ στις πιο σημαντικές πτυχές αυτής της δράσης. Η της πράξη ήταν μία μεταξύ των προτάσεων του Προέδρου Ιούνκερ και της Αντιπροέδρου Μογκερίνη, οι οποίες έλαβαν ομόφωνη υποστήριξη από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη συνεδρίαση στη Σόφια στις 16 Μαΐου, αμέσως μετά την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με ε, το σχέδιο δράσης ε, που αφορά το Ιράν. Αυτή η κατεξιοδότηση κατεξοδότηση πράξη είναι λοιπόν ε, η μεταγραφή μιας ομόφωνης πολιτικής βούλησης. Θα ήθελα να σας πω περί τίνος ακριβώς πρόκειται τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει. Η πράξη ε, σημαίνει ότι το Ιράν θα είναι επιλέξιμη χώρα για την εγγύηση του προπολογισμού που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις, ε, από την ΕΤΕΠ ε, στον εξωτερικό δανεισμό της, κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι η ΕΤΕΠ θα αρχίσει αμέσως να δανείζει στο Ιράν. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι η απόφαση δανειοδότησης και το πού μπορεί μπορεί να δανείσει ή όχι η οχι Παραμένει προνόμιο των ε, ε, αρχών ε, των διοικητικών της ΕΤΕΠ και θα ισχύουν βέβαια όλοι οι κανόνες και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν. Πολύ σημαντική είναι η χρονική στιγμή της πράξης αυτής, η έγκριση της κατεξιοδότηση πράξης στις τον Ιούνιο θα, μπει σε, θα σημαίνει ότι θα μπούμε σε μια περίοδο δύο μηνών στο πλαίσιο της απόφασης ELM. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους κατά τη δίμηνη αυτή περίοδο ή μπορεί να ζητήσουν επιπλέον δύο μήνες ε, για να συσκεφθούν. Όμως η λογική της απόφασης αυτής σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι ότι η πρώτη κύρωση των Ηνωμένων Πολιών θα αρχίσει να ισχύει από τις 6 Αυγούστου. Αν λοιπόν οι δύο μήνες στηριθούν ως προθεσμία, τότε αυτή η αλλαγή ε, είναι ένα σημαντικό ε, ζήτημα αντίδραση σε σχέση με τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε αυτή την ομόφωνη απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και θα αρχίσει να ισχύει μία μέρα πριν από την έναρξη ισχύω ε, της ε, πρώτης ε, ε, ομάδας κυρώσεων των Πολιτειών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λεγμαζιέρ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα προσπαθήσω σε σύντομα να ε, σας κάνω κάποιες προειδοποιήσεις και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μας από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε, για αυτό ε, το γεγονός, ότι είναι πλέον επιλέξιμο δηλαδή το Ιράν ε, Δύο σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, η επιχειρησιακή σημασία είναι πολύ περιορισμένη και δεύτερον, αυτή η απόφαση έχει βαρύτητα για την Ευρώπη μέσω της τράπεζας, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επειδή μπορεί να υπάρχουν σημαντικοί οικονομικοί κίνδυνοι. Καταρχάς, ε, η πολύ μικρή επιχειρησιακή σημασία αυτή της πράξης. Προφανώς ε, η ΕΤΕΠ θα ε, πρέπει να λάβει τις αποφάσεις σε σχέση σχέση με την εφαρμογή αυτής της επιλεξιμότητας και αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί καταρχάς από το Συμβούλιο των Διοικητών ε, ε, θα έπρεπε να υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία για να αρχίσουν ε, οι δραστηριότητε στο Ιράν. Δεν θα μπορέσουν να αρχίσουν αυτέ οι δραστηριότητε αν η ΕΤΕΠ δεν έχει ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει τη ε, με το Ιράν για μια συμφωνία πλαίσιο, επειδή η ΕΤΕΠ είναι υποχρεωμένη να το κάνει με όλε τι χώρε στι οποίε δραστηριοποιείται. Αυτή η συμφωνία πλαίσιο είναι απαραίτητη για να θέτει το νομικό πλαίσιο ε, και ε, τις οικονομικές και χρηματοδοτικές προϋποθέσεις για να μπορέσει η ΕΤΕΠ να προβεί στις δραστηριότητες. Το Ιράν ε, μέχρι σήμερα αποτελεί μια χώρα η οποία δεν σέβεται τους διεθνείς κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος και πράγματι καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνει το σχετικό έλεγχο γιατί το Ιράν είναι μια χώρα στην οποία η ΕΤΕΠ δεν θα έπρεπε τίποτε να χρηματοδοτεί, να χρηματοδοτεί ή πολύ περιορισμένες δράσεις θα έπρεπε να χρηματοδοτεί. Όλα αυτά λοιπόν για το επιχειρησιακό κομμάτι. Όσον αφορά τον οικονομικό κίνδυνο, η τράπεζα χρειάζεται μια καθημερινή πρόσβαση στα, στις διεθνείς κεφάλαια αγορές ε, και συμπεριλαμβάνει βεβαίως και τις αγορές σε δολάρια μέσω των μηχανισμών κυρώσεων ε, δευτερευουσών ε, το να μπορεί η ΕΤΕΠ να θεωρηθεί η ΕΤΕΠ από τις Ηνωμένε Πολιτείε ως οντότητα που βοηθά το Ιράν σημαίνει ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα στους τίτλους ε, που ε, αγοράζει η ΕΤΕΠ σε συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, κάτι το οποίο σημαίνει 10 με 15 δις ευρώ περίπου για προγράμματα της τάξεως των 60 δις η ΕΤΕΠ λοιπόν ε, προβαίνει σε δραστηριότητες ε, σε πολλά νομίσματα. Όλες αυτές θα επηρεαστούν από την ε, επιλεξιμότητα του Ιράν και ειδικότερα σε δολάρια. Ειδικότερα για τα δολάρια μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και να αποδυναμωθεί η ΕΤΕΠ ε, και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο σύνολο των ε, δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ. Θα με ρωτήσετε κατά πόσο όντως έχουν αυτά τα σενάρια επιβεβαιωθεί στις κεφαλαίες Όχι ε, θα έλεγα. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος που ελοχεύει γιατί υπάρχουν επενδυτές εκτός Ευρώπης και μπορούμε να τους ρωτήσουμε ε, κατά πόσο θεωρούν ότι η ΕΤΕΠ πρέπει να επενδύσει στο Ιράν. Υπάρχουν επίσης κάποια άρθρα που απειλούν ευθέως ε, την ΕΤΕΠ ε, στο Wall Street, στη Wall Street Journal που πρόσκειται πολύ στον πρόεδρο και υπήρξαν πολύ εχθρικά δημοσιεύματα όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την αποφασή της και η ΕΤΕΠ παρεμποδίστηκε την, ε, ε, στη δυνατότητα έκδοσης ενός δανείου, κάτι το οποίο δεν έγινε και έτσι έκλεισε το παράθυρο ε, της αγοράς που επέτρεπε αυτήν την δανειοδότηση και δεν ξανά άνοιξε αυτό το παράθυρο. Αυτό οδηγεί την ΕΤΕΠ να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την απόφαση αυτή, ότι είναι επικίνδυνη και ότι τουλάχιστον θα μπορούσαμε να περιμένουμε να γνωρίζουμε καλύτερα το πεδίο των ε, κυρώσεων ε, και των μέτρων ε, των Ηνωμένων Πολιτειών πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε. Λοιπόν, τώρα... Είμαστε σε επίπεδο στρατηγικής σκέψης και αντιπαράθεσης ανάμεσα στην πολιτική βούληση από τη μία και τις στάσεις των αγορών από την άλλη. Να δούμε αν το ευρώ κάποτε γίνει πολεμικό όπλο στον τομέα των εμπορικών. Monsieur Fleckenstein, qui est rapporteur permanent pour l'Iran à la Commission des Affaires étrangères, car euh, Monsieur le rapporteur. Λοιπόν, ο κύριος Φλέκενστάιν, ο εισηγητής ε, θα πρέπει να φύγει στις 11, είναι 11, γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα. I, uh, Ε, μπορεί να μείνω και λίγο παραπάνω. Μια ερώτηση έχω μόνο. Μας προειδοποιήσατε. Για τις απόψεις της τράπεζας για το θέμα αυτό, της ΕΤΕΠ, έχω μια ερώτηση. Καλύτερη εναλλακτική λύση έχετε να μας προτείνετε. Τι θα μας προτείνετε να κάνουμε εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Στον κύριο de Mazière, την απευθύνετε την ερώτηση, ο οποίος θα σας απαντήσει τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως σας είπα, επιχειρησιακά, λειτουργικά δεν θα έχει πολύ μεγάλη παρουσία στο Ιράν. Α, ξέχασα να αναφέρω ότι είναι και πολύ μικρό το περιθώριο το δημοσιονομικό και το οικονομικό που έχουμε για την εξωτερική εντολή. Είναι αρκετά περιορισμένη λοιπόν η δράση ε, της τράπεζας στο Ιράν. Γιατί θα εκτεθεί σε κίνδυνο και η ίδια και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στις κεφαλαιογορές σε δολάρια. Η εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι να βρεθεί ένας πιο σύντομος τρόπος να είναι σε άμεση σχέση τα ευρωπαϊκά οικονομικά με το Ιράν, με, χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τη σύσταση ενός καταπιστευματικού ταμείου μια πρόταση είναι αυτή. Ομολογώ ότι δεν έχω μελετήσει σε βάθος ε, τις ε, διάφορες δυνατότητες. Ε, κύριε Σιγητά τη επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Σα εμπνέει αυτή η απάντηση, κάποια αντίδραση, πλέον κάποια σκέψη, Ωραία, θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεβαντόφσκι, που είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ιράν. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της αντιπροσωπείας ε, ε, ε, πρέπει να πω ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν ήταν μια επιτυχία της πολυμερού συνεργασίας στον κόσμο και η καταγγελία της ε, είναι πολύ αρνητική. Το θέμα δεν ήταν αυτή, αυτή η συμφωνία για τα πυρηνικά, ήταν ε, το άνοιγμα της χώρας, η ενίσχυση των προοδευτικών δυνάμεων και των δημοκρατικών και η δυνατότητα να ασχοληθούμε με θέματα όπως είναι και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατάστασή του στο Ιράν. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν είναι ευρύτερη εικόνα. Από την αρχή λοιπόν το πρόβλημα ήταν οι τράπεζες και τα οικονομικά για το ε, ε, οικονομικό αυτό μέρισμα υπέρ των ανθρώπων στο Ιράν. Τώρα η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη. Η ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή είναι σαφέστατη και την έχουν επικυρώσει εγκρίνει ε, όλοι οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σόφια για την ασφάλειά μας και την παγκόσμια ασφάλεια και τη στρατηγική μη διάδοση των πυρηνικών. Άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, το νόμιμο εμπόριο με το Ιράν. Και εδώ χρειαζόμαστε δύο κατεξοδότηση πράξεις. Η μία ε, για αναβάθμιση ε, της ε, σχέσεις και το δεύτερο είναι η δράση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων η οποία έχει τους λόγους της προφανώς να είναι προσεκτική και επιφλακτική αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αν θέλουμε εμείς να ανταποκριθούμε στο δικό μας σκέλος της συμφωνίας η οποία για μας συνεχίζεται. Προσωπικά πιστεύω ότι η απόφασή μας ε, είναι και επίδειξη οικονομικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ε, και την ε, εγκρίνω και την προσωπογράφω εξονόμως της Ιρανικής Αντιπροσωπείας για το Ιράν. Ευχαριστώ. Είπατε ότι οι μέτοχοι της τράπεζας θα το επιθυμούσαν. Όμως η ίδια η τράπεζα δυσκολεύεται να εφαρμόσει την ομόφωνη επιθυμία των μετόχων της η μόνιμη εισηγήτρια για τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, η κυρία Γουάρδια Σάμπαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να διευκρινίσω εγώ ειδικά τίποτα. Μιλάμε για επενδύσεις στο Ιράν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην ουσία κάνουμε μία κίνηση σε επίπεδο διπλωματικό, μία πρόταση ε, στα πλαίσια της συμφωνίας και στα πλαίσια της απειλής των ε, κυρώσεων από πλευράς ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μια διπλωματική κίνηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυρίας Μογκερίνη είναι κάτι το πιο σημαντικό από τις μελλοντικές οικονομικές ή χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις. Προφανώς το Διοικητικό Συμβούλιο ε, της Τράπεζας Επενδύσεων είναι εκπρόσωποι των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι ίδιες αυτές χώρες αποφάσισαν να γίνει αυτό το διπλωματικό άνοιγμα, αυτή η διπλωματική κίνηση προς το Ιράν. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να δούμε τι συνέπειες θα έχει κάτι τέτοιο ε, για την πρόσβαση στην χρηματοδότηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες από πλευράς της τράπεζας για τις πιθανές επιπτώσεις στην χρηματοδότησή της από ένα τέτοιο μέτρο, από μια τέτοια κίνηση. Προς το παρόν νομίζω ότι οι αποφάσεις μέχρι τώρα και η πολιτική βούληση είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό από μόνο του. Και η συμπερίληψη του Ιράν στις ε, σε εισαγωγικά επενδύσιμες χώρες ε, δεν σημαίνει ότι θα γίνουν επενδύσεις. Ε, πάντα έτσι και αλλιώ για επενδύσεις σε τρίτες χώρες απαιτείται η ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα και προσοχή. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ είναι να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, για μια πολιτική κίνηση, για ένα διπλωματικό διάβημα. Ίσως κάποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το δικό της νόμισμα, το ευρώ, σαν μέσο άμυνας οικονομικής και εμπορικής πολιτικής όπως και το κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό θα έχει νομίζω νόημα. Σαρβάμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας ότι ναι μεν δεν γνωρίζουμε τις τεχνικές συνέπειες και τις χρηματοπιστωτικές συνέπειες ε, της χρήσης των κοινοτικών πιστώσεων, οι συνέπειες ε, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι κάτι που θα πρέπει να ε, εξεταστεί και να εκτιμηθεί. Δεν θα πρέπει να πιστεύουμε πιστεύει όμως κάποιος ότι υπάρχει απόλυτη μειοφωνία για τέτοιου είδους επενδυτικές δραστηριότητες. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε λίγο τη στρατηγική του κυρίου Φλέκενστάιν και να μην περιμένουμε μία επιπλέον απάντηση αλλά να εκφράσουμε την άποψή μας. Εμείς έχουμε πάρει κάποιες ξεκάθαρες θέσεις για την ιδέα της ιστορικής αυτής συμφωνίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα και φέρον της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το αμφισβητήσουμε αυτό, ελπίζω να έχουμε κάνει το σωστό, θα το δείξει αυτό στο μέλλον, αλλά δεν χρειάζεται να βιαστούμε, το Ιράν έχει χρήματα, έχει πόρους, αλλά το πώς τους χρησιμοποιεί δεν μπορεί να δώσει το καλό παράδειγμα. Είναι αντίθετα αυτά που κάνει με όλα αυτά τα οποία εμείς επιθυμούμε και προκρίνουμε. Είναι αντίθετα λοιπόν αυτά τα οποία πράττει η χώρα αυτή σε σχέση με τις δικές μας αρχές. Τώρα ξαφνικά το να αρχίσουμε να στέλνουμε χρήματα σε κάποιες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μεταρρυθμιστές, είναι μια δικτατορία η οποία με ε, ιδιαίτερη βία ε, καταστέλει τις διεκδικήσεις των λαών της ε, και παρεμβαίνει αρνητικά στην περιοχή και στη Μέση Ανατολή. Η στρατηγική της δεν είναι, του Ιράν ενώ, δεν είναι μια στρατηγική ειρήνης. Ευχαριστώ κύριε Σάρφαμα. Ήταν ο πρώτος από έναν κατάλογο ομιλητών της Επιτροπής Προϋπολογισμών ή και της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σιουατάγνιο που αντικαθιστά τον κύριο Φλίντς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Κύριε Άγνιο, έχετε το λόγο. Το να καταστήσουμε επιλέξιμο το Ιράν είναι για οικονομική στήριξη, είναι κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Εγώ σαν βουλευτής του UKIP είμαι κατά της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων και των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε τρίτες χώρες. Αυτό θα δημιουργήσει πολιτικό και διπλωματικό πρόβλημα για το Ιράν. Ξέρω όμω γιατί το κάνετε αυτό ε, ακριβώς μέσω της πυρηνικής συμφωνίας, της συμφωνίας για τα πυρηνικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι θα ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή εις βάρος της αμερικανικής ισχύως. Ε, αν αποχωρήσουν τώρα οι Αμερικανοί, πώς αυτό θα επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα μιας και χρησιμοποιεί τις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές αγορές για να δανειστεί χρήματα η τράπεζα λοιπόν δεν είναι ευτυχής για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί παίρνει χρήματα από τις Αμερικανικές αγορές, χρήματα αγορές. Έτσι κι αλλιώς πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ που έχουμε έτσι κι αλλιώς μαζί του πολλά προβλήματα. Και νομίζω ότι το Ιράν προετοιμάζεται για να αποτύχει η συμφωνία. Ο υπεύθυνο Ιρανός εκπρόσωπος είπε ότι θέλουν να δημιουργήσουν νέες τεχνικές μονάδες για την επεξεργασία καυσίμων. Συνεπώς λοιπόν η κατεξουσιοδότηση πράξη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δημοκρατική πρόταση για ένα τόσο περίπλοκο θέμα και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ψηφοφορία αν δεν εκφράσει αντίρρηση το Κοινοβούλιο και απλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά την επανεισαγωγή των κυρώσεων. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να εκφράσουμε την αντίρρησή μας, θα πρέπει να το κάνουμε το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεπρέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Δεν θα μιλήσω επί της ε, ουσίας ε, της απόφασης, αλλά ε, θα επικεντρωθώ κυρίω στι πολιτικέ συνέπειε που μπορεί να έχει. Είναι γεγονό ότι στο πλαίσιο τη τρέχουσα συγκυρία δεν θα μπορούσε να ειδωθεί ω αντιαμερικανική πράξη. δεν θα μπορούσε παρά να θεωρηθεί αντιαμερικανική πράξη. Ε, δεν έχω όμω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό, όμως θα θεωρηθεί ε, ως πράξη υποστήριξης ε, ε, των ε, Ιρανικών αρχών. Είναι μια θεοκρατική δικτατορία η οποία ε, αποσταρτεροποιεί τις διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, ε, της ε, Συρίας, της Ιεμένης και το να κάνουμε μια οποιαδήποτε πολιτική κίνηση ανεξαρτήτως της απόφασης και της άποψης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αποτελεί μια υποστήριξη αυτού του καθεστώτος. Λοιπόν, το πρώτο ε, στοιχείο που υπόθηκε, η μία πιθανότητα, είναι μία εντελώς θεωρητική απόφαση η οποία δεν θα ισχύσει. Άκουσε αυτό που μας είπε η ΕΤΕΠ. Ε, θεωρητικά ε, μπορεί να υπάρχει πιθανότητα, αλλά σε στην πράξη μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Ε, άρα, άρα τι νόημα έχει. Αν εφαρμοστεί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Θα μπορούσε δηλαδή για παράδειγμα να έχει έναν αντίκτυπο για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις δραστηριότητες της ΕΤΕΠ. Γι' αυτό προτείνω εμείς στην Επιτροπή μας, ε, που είμαστε Επιτροπή Προϋπολογισμών, να αντιδράσουμε αν αυτή η απόφαση ληφθεί και αν εφαρμοστεί, θα ε, πρέπει να υπάρξει μία αξιολόγηση επιπτώσεων. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε το ή άλλως, κάνουμε και για τα υπόλοιπα θέματα. Και εδώ μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ε, αν όντως εφαρμοστεί η απόφαση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν επισήμως να ζητήσω η Επιτροπή Προϋπολογισμών να ζητήσει μία μελέτη επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΤΕΠ για να μας εξηγήσει ακριβώ ποιοι θα είναι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και επίση να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεδομένη της θέσης του κυρίου Τραμπ, ε, ποια είναι τα μέτρα που θα λάβει για την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θα συνεχίσουν ε, να δραστηριοποιούνται στο Ιράν, γιατί μέχρι τώρα άκουσα διάφορες δηλώσεις, αλλά δεν είδα κανένα ε, επιχειρησιακό μέτρο, οπότε θα ήθελα να ζητήσουμε μία μελέτη επιπτώσεων πριν από ε, την απόφαση αυτή. Πρόεδρο. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μούρεσαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης ηγετής του ΕΛΚ για το θέμα αυτό, έχω να πω τα εξής. Πρώτον, είναι δημοκρατία το Ιράν που να σέβεται τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως και τα κράτη μέλη. Απάντηση όχι, προφανώς. Ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε και συμφωνώ με τα όσα είπε ο Ζεράρ Ντεβρέ και ο κύριος Σαρβάμα προηγουμένως για την κατάσταση στο Ιράν. Ωστόσο, υπήρξε πολιτική συμφωνία σε επίπεδο συμβουλίου με όλα τα κράτη-μέλη μας που ε, λέγει ότι είμαστε τμήμα αυτής της συμφωνίας για τα πυρηνικά. Και διάφορες εξελίξεις λέγουν ε, ότι μια συμφωνία αυτή με ένα καθεστώς που δεν μας αρέσει και από ό,τι φαίνεται δεν τους αρέσουμε κι εμείς, η συμφωνία όμως ε, λειτουργεί. Και μα λένε και οι ειδικοί εμπειρογνώμονε μα εδώ του Κοινοβουλίου για θέματα εξωτερική πολιτική ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτή τη συμφωνία παρά τη μονομερή ε, απόφαση του σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ. Για να τη διαφυλάξουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία η πρόταση τώρα επιτάπητο είναι να εγγραφεί το Ιράν στον κατάλογο επιλέξιμων κρατών. Αυτό τι σημαίνει. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα χρηματοδοτούμε έργα στη χώρα και η Ρωσία είναι στον κατάλογο των επιλέξιμων κρατών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν έχει παρουσία από το 2015 με δανειοδότηση, αν δεν απατώμε στη Ρωσία. Γι' αυτό λέγω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτή την κατεξουδότηση πράξη, να επιτρέψουμε να συμπελευθεί στον κατάλογο επιλέξιμων χωρών το Ιράν, γνωρίζοντας ότι έχουμε την πολιτική δέσμευση Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συμμετέχει σε έργα που ανταποκρίνονται στους δικούς της στόχους και σε καμία περίπτωση δεν θα καταλήξουν στα χέρια του καθεστώτος για να τα χρησιμοποιήσει για αλότριους ε, σκοπούς προς τους δικούς μας. Αυτή είναι η απόφαση. Η ΕΤΕΠ είναι τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οφείλει να ε, υλοποιεί τι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουμε εμεί τα τρία θεσμικά όργανα. Βεβαίως, πάντα ελαχιστοποιώντα του κινδύνου. Και με όλη τη συμπάθεια που έχω προ την ΕΤΕΠ και οι συνάδελφοι τη ΕΤΕΠ ξέρουν πόσο εκτιμώ το έργο του και τη συνεισφορά του σε σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, όσο και να αγαπώ την ΕΤΕΠ, ο ρόλο της είναι να υλοποιεί τι αποφάσεις που λαμβάνουν ε, σε πολιτικό επίπεδο τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ναι, αν είναι αυτή η πολιτική θα πρέπει να υλοποιείται κιόλα. Ε, παρέθεσε ο εκπρόσωπο τη ΕΤΕΠ ένα άρθρο της Wall Street Journal που με τη σειρά του αναφέρει κάποιε πηγές του Λευκού Οίκου για τους κινδύνους στην Αμερικανική αγορά και με όλο το σεβασμό για την εφημερίδα αυτή, εμείς πρέπει να πάρουμε εδώ πολιτικές αποφάσεις και να μην βασιζόμαστε σε δημοσιεύματα που ε, παραθέτουν πηγές του Λευκού Οίκου. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμείς Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε, αποκλίνουν στη συμφωνία με το Ιράν από εκείνους του Λευκού Οίκου. και επιθέσεις ε, ακούσαμε και το ΙΤ κυκλοφόρησαν προς την κατεύθυνσή μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να πάρουμε μια απόφαση. Και δεν χρειάζεται απαραίτητο να απαντούμε σε πιέσει, ακόμα και σε απειλέ που εκτοξεύονται και δημοσιοποιούνται και από το μέσο που παραθέσατε. Προσοχή λοιπόν, με τρόπο συγκρατημένο και υπεύθυνο να μην αντιταχθούμε σε αυτή την κατεξοδότηση πράξη, να παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις. Άκουσα πολύ προσεκτικά και τα όσα είπε ο Ζεγά. Και να παρακολουθούμε και τι κάνει η ΤΕΠ στο Ιράν. Να είμαστε σίγουροι ότι φυγερμαζόνται με τους δικούς μας στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Κόλμελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απολύτω με τα όσα άκουσα από του συναδέλφου. Θέλω όμω να τονίσω κάτι ακόμα ρητά. Κατά κανόνα θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση όπω και στο παρελθόν. Ποιο είναι το πολιτικό υπόβαθρο και τι ζητάνε από εμά Επιτροπή Προπολογισμών. Είναι γνωστά τα πολιτικά, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε όλα όσα υπόθηκαν ήδη. Αλλά δεν είναι δική μα δουλειά αυτό. Η δική μα δουλειά ποια είναι, να καθίσουμε να σκεφτούμε τώρα τα μέτρα που προτείνονται μέσω της ΕΤΕΠ να εγγυηθούμε χρηματοδοτήσεις είναι ο σωστός φορέας για να κάνουμε μια πολιτική κίνηση που είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Και εκεί άκουσα πάρα πολύ λίγα ειλικρινά που να συνηγορούν προς την κατεύθυνση αυτή και άκουσα μερικά που είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτά που λέει η ίδια λοιπόν η ΕΤΕΠ. Άρα προσοχή και προεδοποιώ. Επειδή έχουμε μια πολιτική τώρα ε, εξωτερική μην χρησιμοποιήσουμε το λάθος εργαλείο που θα έχει αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί θα είναι για άλλη μια φορά αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία τα πολιτικά, τα έχουμε συμφωνήσει, ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ ωραία και να το υποστηρίξουμε, αλλά να βρούμε και το σωστό τρόπο και τα σωστά μέτρα να το κάνουμε αυτό. Και προς το παρόν είναι μάλλον περισσότερα τα ερωτηματικά παρά οι απαντήσεις. Um, Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εμένα μου φαίνεται πολύ ε, περίεργο ότι ο τρόπος με τον οποίο οι όροι με τους οποίους μιλούμε για την πυρηνική συμφωνία ε, του Ιράν που λέμε ότι η συμφωνία θα έπρεπε να ε, πηγαίνει πολύ παραπέρα από ε, τον έλεγχο της ανάπτυξης και της μη διασποράς των μέσων μαζικής καταστροφής στο πλαίσιο ε, των συμφωνιών που έχουν γίνει για την ε, εξαγωγή των όπλων και τον έλεγχο των εξαγών όπλων, πάντοτε υπήρχαν συμφωνίες από το Δεύτερο Παγκόσμιο ε, Πόλεμο και εξής. Δεν πιστεύω ότι το, η πυρηνική συμφωνία του Ιράν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το καθεστώς, να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνεχίσει να κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε χτες, για παράδειγμα, ε, κρέμασε έναν ε, προφανώς αθώο άνθρωπο ε, αυτά δεν είναι κάτι, δεν είναι πράγματα τα οποία τα ενέκρινε σε καμία περίπτωση μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Επίσης είναι και περίεργη στρατηγική σκέψη να λέει κανείς ότι είναι μια πολύ καλή χρονική στιγμή να λάβουμε μια απόφαση. Σήμερα ακούσαμε ε, από διάφορα ε, μέλη αλλά και αξιωματούχους οι οποίοι μας ε, ανέφεραν όλες αυτές τις πτυχές. Δεν είναι καθόλου σαφές το παιχνίδι αυτό και όταν κανεί μπαίνει στη διαδικασία να λαμβάνει αποφάσει που δεν χρειάζεται να ληφθούν για λόγου μια κίνηση, ε, έχει πλέον εγκαταλείψει ε, το ρεαλισμό και τη στρατηγική σκέψη επίση. Οπότε δεν ξέρουμε τι συνέπειε, δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι επόμενε πολιτικέ εξελίξει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, διαφωνίε όσον αφορά τους κινδύνου και δεν γνωρίζουμε ακριβώς ε, ποια θα είναι η αντίληψη, δηλαδή πώς θα ε, γίνουν αντιληπτές αυτές οι αποφάσεις, ούτε τις συνέπειες αυτών. Ε, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπούμε σε καμία συμφωνία που θα μας υποχρεώσει να δανείσουμε χρήματα ε, σύντομα. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση και δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς ε, ποιες διαδικασίες ισχύουν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να μπαίνουμε σε μια διαδικασία κατά την οποία παίρνουμε μια απόφαση επειδή μας φαίνεται ότι επί της αρχής είναι καλή ιδέα να πάρουμε μια απόφαση χωρίς να σκεφτόμαστε ρεαλιστικά και δεν νομίζω ότι οι διεθνείς σχέσεις λειτουργούν έτσι. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν εξετάζουμε μια τέτοια απόφαση πρέπει να σκεφτούμε ε, κατά πόσο υπάρχει μια διαφωνία όχι μόνο όσον αφορά την απόφαση επί της αρχής αλλά και σε σχέση με το χρονισμό αυτής της απόφασης που δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουκνερ από την Επιτροπή Εξωτερικών. Μπουκνερ. Ναι. Πιστεύω ότι εδώ δεν θα πρέπει να συγχαίουμε διάφορα πράγματα που ακούστηκαν στη συζήτηση ανανεμιγμένα. Από τη μια έχουμε τη συμφωνία για τα πυρηνικά και τον αφοπλισμό. Λόγω του αφοπλισμού ή λόγω των εξοπλισμών υπήρξαν κυρώσεις. Τώρα υπάρχει άλλο θέμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν εκεί υπήρχαν διαφορετικές κυρώσεις, ξεχωριστές, οι οποίες δεν θίγονται, παραμένουν, δεν έχουν αρθεί. Μετά υπάρχει το πρόβλημα της συμμετοχής ε, και της εμπλοκής του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Και εκεί ε, είναι κάτι που δεν μας αφορά αυτό. Το μόνο που μας απασχολεί τώρα είναι η συμφωνία για τα πυρηνικά. Για ποιο λόγο το Ιράν προχώρησε στη σύναψη αυτή τη συμφωνία. Εγώ, ξέρετε, είμαι πυρηνικό φυσικός. Μπορεί να είμαι και μοναδικός στο Κοινοβούλιο. Εγώ δεν θα την υπέγραφα αυτή τη συμφωνία. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει στην παραγωγή ε, πυρηνικού υλικού για ειρηνική ε, χρήση. Ε, σταματάνε τον εμπλουτισμό του ουρανίου τώρα σε ένα επίπεδο που εγώ προσωπικά δεν θα το είχα δεχτεί. Εντάξει, τώρα το Ιράν το δέχτηκε. Υπέγραψε ακριβώς διότι ο, ο λαός κυρίως ήλπιζε βελτίωση του βιωτικού του επίπεδου. Και αυτό είναι το κλειδί. Ε, το Ιράν ήδη από τώρα έχει πει ότι θα συνεχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο εάν καταρρεύσει αυτή η συμφωνία. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα έχουμε πυρηνικού εξοπλισμού ή όχι. Εάν όχι, χρειάζεται και ο λαό ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα είναι επενδύσεις δικές μας. Εάν καταρρεύσει η συμφωνία αυτή, τότε η Σαουδική Αραβία ήδη από τώρα έχει δηλώσει ότι θα αποκτήσουν και η ατομική βόμβα και είναι λεωφόρο αυτή που ανοίγεται μπροστά τη για να το κάνει αυτό. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Και αν αποκτήσει πυρηνική βόμβα και η Σαουδική Αραβία έπονται και άλλοι εθελοντές. Κάποιοι που έχουν ήδη βόμβα. Εγώ ήμουνα ε, στη Νέα Υόρκη το 2015 στη διάσκεψη για τη μη διάδοση και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ σαφής. Λοιπόν, έχουμε τώρα ακριβώς αυτή την επιλογή. Θα τηρήσουμε τη συμφωνία αυτή με το Ιράν για τα πυρηνικά. Με τη δυνατότητα άρση των κυρώσεων που συνδέονται με αυτές. Ή θα αφήσουμε ε, αυτή τη ξέφρενη πυρηνική κούρσα στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ερώτημα και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε και δεν θα πρέπει να μας εμποδίσουν λίγα χρήματα να το κάνουμε αυτό. Ήταν πολύ επίπονος ο δρόμος μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την εμπειρογνωμοσύνη σας μαζί μας. κυρία Λαλόντ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο ότι πρέπει δηλαδή να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Νομίζω ότι ο κίνδυνος ε, του να μην σεβαστούμε κατά γράμμα τη συμφωνία αυτή είναι πολύ υψηλότερος ε, από το να μην τη σεβαστούμε. Η Σαουδική Αραβία ούτω ή άλλω είναι απολύτω έτοιμη να αναπτύξει την ατομική βόμβα αν ε, το Ιράν ξαναμπεί στην ε, πυρηνική κούσα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για όλη την περιοχή. Γνωρίζω λιγάκι το Ιράν. Μπορώ ε, να ε, σας πω ότι ό,τι κύρωση έχουμε επιβάλει στο Ιράν, ο Ιρανικός λαός το, την υφίσταται. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που επιβάλλουμε κυρώσεις. Ο λαός είναι αυτός που τις υφίσταται και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ κακό πολιτικό μήνυμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην σεβαστεί ε, πλήρως αυτήν την ε, συμφωνία με το Ιράν. Ζεράρ, τι λες ακριβώς. Μα δεν είναι αυτό το θέμα, λέει ο κύριος Δεπρέ ε, εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά είμαι με τη διατήρηση της συμφωνίας δεν σημαίνει ότι θα περάσει το Ιράν από το ένα κατάλογο στον άλλον. Ε, ε το, ε, δεν σημαίνει αυτό ότι διακυβεύουμε την ε, αποφασιστικότητά μας και την αφοσίωσή μας στην πυρηνική συμφωνία. Ναι, εντάξει, αλλά ένα τμήμα της συμφωνίας αφορά ακριβώς το ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να επενδύσουν στο Ιράν. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι μηχανισμοί ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να ε, επενδύσουν. Η Total φεύγει σιγά σιγά και άλλες επιχειρήσεις φεύγουν, ε, συνεπώς θα είναι και η Πεζό, επίσης. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν ε, και δεν ξέρω λοιπόν ε, ποιο είναι το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ενδιαφέρει και ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας σε όλη αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι δεν έχουμε και πολλά να κερδίσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανένα άλλος να πάρει το λόγο. Ούτω ή άλλω αυτό το θέμα δίνει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους να αξιολογήσουν την πολιτική του ισχύ ε, Ο κύριος ε, Ντεπρέ μας ε, είπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, την αξιολόγηση κινδύνου και τις αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσαν να υπάρξουν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αν μαζικά επενδύσει στο Ιράν να ολοκληρώσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική και ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε στον εκπρόσωπο της ΑΕΕ, e τον κύριο Τόρστεν ε, Μπάρφρεντ, να μας ε, πει και εκείνος ε, την άποψή μας, την άποψή του. Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχει υποθεί και προηγουμένως από κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου ότι υπάρχει γενικό συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της πυρηνικής ε, συμφωνίας, ε, ακόμη και αν δεν συμμετέχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η ανακούφιση των κυρώσεων σημαίνει ότι θα συνεχίσει μια οικονομική συνεργασία με το Ιράν και αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα της συμφωνία. οπότε οποιαδήποτε μέτρα μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο, υποστηρίζουν και τη συμφωνία μακροπρόθεσμα. Ε, όσον αφορά τώρα το τρέχον γεωπολιτικό ε, κλίμα, δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ε, πώς έχουν τα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό το μέτρο που υπάρχει, υπάρχουν και άλλα μέτρα. Προσπαθούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Υπάρχουν μέτρα που προσπαθούμε να συζητήσουμε και με τα κράτη-μέλη και για να δούμε πώς μπορούν να συνεχίσουν οι εισαγωγές πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη νέα κατάσταση, ε, αν υπάρξουν ε, επιπλέον αμερικανικές κυρώσεις. Πάντως, ε, εμείς υποστηρίζουμε τη, την ε, συνέχιση της συνεργασίας με το Ιράν, όπως δήλωσε και το Συμβούλιο Εξωτερικών το 2016. Υποστηρίζουμε, λοιπόν, τα μέτρα αυτά. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Προτείνω λοιπόν να το κλείσουμε εδώ. Το θέμα αυτό, οι συντονιστές στην επόμενη συναντρίασή τους θα αποφασίσουν, μάλλον με την, όχι την, την επόμενη, είναι πήγον, μάλλον με τη γραπτή διαδικασία θα αποφασίσουν αν χρειαστεί να ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας πρόταση αντίρρησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. κάθε πολιτική ομάδα, μια πολιτική ομάδα ή 40 βουλευτές μπορούν να καταθέσουν στην Ολομέλεια βάσει του άρθρου 105 του κανονισμού εντός των γνωστών προθεσμιών αυτή την, το αίτημα. Σε ό,τι αφορά όμως την Επιτροπή Προϋπολογισμών, η πρόταση αντίρρησης θα πρέπει να είναι αντικείμενο αξιολόγησης, εκτίμησης και απόφασης των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Και βλέπουμε ποιο είναι το δυναμικό της ίδιας πολιτικής ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα χρειαστεί μάλλον κάποια συζήτηση, γιατί όταν οι Αμερικανοί χάρη στο δολάριο μπορεί να επιβάλλουν βαρύτατα πρόστιμα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή και ευρωπαϊκές τράπεζες, ποιο είναι ε, το όραμα ή η θεώρηση της Ευρώπης απέναντι σε όλα αυτά. Μπορούμε να φανταστούμε κάποια στιγμή το ευρώ να έχει την ίδια θέση που έχει διεθνώς το δολάριο και τι σημαίνει το δολάριο για τις Αμερικανικές αρχές θα σημαίνει το ίδιο και το ευρώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές και τους συναδέλφους της Επιτροπής Εξωτερικών, τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΤΕΠ και της ΑΕΔ. Λήξη στη συζήτηση αυτή για σήμερα το πρωί και παίρνουμε στο επόμενο θέμα που είναι η εντολή της Επιτροπής Προπολογισμών στους εκπροσώπους της για το τριμερή διάλογο για μια πρώτη αντίδραση του Κοινοβουλίου για το σχέδιο προπολογισμού 2019. Θα δώσω μέσα το λόγο ε, στον εισηγητή μας, τον γενικό εισηγητή, τον κύριο Ντανιέλε Βιώτη. Θυμίζω ότι θα πρέπει να τελειώσουμε οπωσδήποτε στις 12.30. Grazie Presidente, ehm, Ευχαριστώ συνάδελφε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είδαμε την πρόταση προϋπολογισμού α, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και την πρόταση για την εντολή για τον τριμερή διάλογο ο οποίος θα πρέπει να, η οποία θα πρέπει μάλλον να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του μηνός Ιουλίου. Εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό ε, έναν βαρετό και τεχνικό κατάλογο των βασικών χαρακτηριστικών της πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν θα είμαι ιδιαίτερα πολιτικός και θα σταθώ στα περισσότερα τεχνικά θέματα θέση προς θέση. Από το 1α 9% αύξηση στι πιστώσει σε σχέση με το 18, πιστώσει υποχρεώσεων σε σχέση με το 18. Εδώ εκφράζουμε την ικανοποίησή μας και για ε, την ενδυνάμωση του ΕΦΣΥ και για την πρωτοβουλία της άμυνας, αλλά δεν θα πρέπει να πηγαίνει σε προγράμματα τα οποία έχουν ήδη σημειώσει μια κάποια επιτυχία θα πρέπει επίσης να διατηρήσουμε τα προγράμματα αυτά και να αυξήσουμε επίσης τα προγράμματα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία μας, την ευρωπαϊκή οικονομία, τις επιχειρήσεις μας, τα πανεπιστήμια μας, τις ε, δημόσιες διοικήσεις μας όπως το ΙΡΑΖ, το Horizon 2020. Τώρα, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας εδώ και την ικανοποίησή μας που ξεκίνησε επιτέλους το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι αποδεκτό να αφήνει στις αρμόδιες επί του προπολογισμού αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευθύνη να βρουν τις απαιτούμενε πιστώσει. Πρέπει να το κάνει αυτό η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κάνει τις απαιτούμενε προβλέψεις. Για το 1β, αύξηση 8% σε σχέση με το 18%. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι τα προγράμματα του πολιετούς δημοσιονομικού και οι καθυστερημένες πληρωμές έχουν μειωθεί με πολύ σημαντικό τρόπο. Σχετικά τώρα με το κύριο τμήμα του 1β, Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τους νέους, διατηρείται και ενισχύεται. Αν και τροποποιείται η συμφωνία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίδει εγγυήσεις για το επίπεδο των χρηματοδοτήσεων. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει το 1Β αυτό στο μέλλον και στα πλαίσια της τελικής συμφωνίας με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Για το 2 προβλέπεται μία αύξηση 1,2% για το 3 σημαντική αύξηση 7,7 σε σχέση με το 2018. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας εδώ για θέματα όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση. Δεν μπορούμε όμως να ξεχνάμε και το υπενθυμίζουμε στην έκθεση ότι η αύξηση αυτή ε, ακολουθεί μετά από πολλαπλές μειώσεις και περικοπές τα προηγούμενα χρόνια Συνεπώς λοιπόν η πραγματική αύξηση δεν ξεπερνά το 2%. Αυτές είναι οι ουρά θα έλεγα οι συνέπειες ε, της ε, μεταναστευτικής κρίσης. Για τέταρτη χρονική ε, περίοδο στο 3 υπάρχει πλήρης εξάντληση των δυνατοτήτων και δεν έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε πιθανά απρόβλεπτα συμβάντα. Να θυμίσουμε ότι τίποτα δεν θα έχει καθοριστεί αν δεν υπάρξουν αποφάσεις ε, ταχύτατα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Γι' αυτό μιλάμε, αν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, θα πρέπει επίσης να υπάρξει ενίσχυση των δυνατοτήτων συνεργασίας και συντονισμού των διοκτικών αρχών. Στο 4 υπάρχει και εδώ σημαντική αύξηση. Αυτό όμως συνδέεται κυρίως, δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις, με το δεύτερο τμήμα της χρηματοδότησης της Τουρκίας για τους πρόσφυγες. Περί αυτού πρόκειται. Ε, είναι ικανοποιητική έτσι και αλλιώς η αύξηση βέβαια. Κινητοποιείται πλήρως το περιθώριο βέβαια και δεν αφήνεται κανένα περιθώριο στο τέταρτο ε, για άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είναι απαραίτητα. Ε, επίσης και τα 100 εκατομμύρια για τη Μεσόγειο είναι κάτι το οποίο δεχόμαστε αλλά δεν είναι το ύψος της ικανοποιητικό για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις τώρα σε συνεργασία με τους συναδέλφους εμείς εδώ θα παρακολουθήσουμε αν θέλετε και θα χρησιμοποιήσουμε τον τεχνικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση συγκεκριμένα πολιτικά κριτήρια τα οποία η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα χρησιμοποιήσει. Σας ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Θα περάσουμε τώρα στους Χολ Χολμέιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συνάδελφο Βιώτη για την εξαιρετική του έκθεση. Με τις κατευθυντήριες γραμμές ορίζονται κάποιες προτεραιότητες οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά υπάρχουν και κάποια προβλήματα για κάποιες δυσκολίες που ανέφερε ο κ. Βιώτη, ε, η βοήθεια για τη γειτονία, αναπτυξιακή βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια, όπου οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις, να αποσοβήσουμε κρίσεις, να βοηθήσουμε ανθρώπους στην Αφρική και σε άλλες περιφέρειες. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και θα χρειαστούμε στο μέλλον για το σκοπό αυτό. Οπότε βλέπω λίγο επικριτικά το γεγονός ότι η Κομισιόν ζητάει από εμά περισσότερα χρήματα για την ε, Τουρκία, ενώ τα κράτη-μέλη αποφεύγουν να δεσμευθούν. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία, αλλά δεν μπορούμε αδιαλείπτως να ηθικολογούμε και να βγάζουμε διάφορα ε, ωραία κηρύγματα, αλλά όταν πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια, για ε, βοήθεια αναπτυξιακή και μέτρα για να βοηθήσουμε τις περιφέρειες να σταθεροποιηθούν, τότε να μην ακολουθούν οι πληρωμές. Διότι υπάρχουν συμφωνίες με κάποια κράτη που χωλένουν στην υλοποίησή τους, είναι πάρα πολύ διστακτικές και επιφυλακτικές όταν υλοποιούνται. Γι' αυτό και ο κόσμος φεύγει από τις χώρες του και έρχεται εδώ γιατί δεν έχει υποστήριξη ή τουλάχιστον επαρκή υποστήριξη. Να πω και μερικά ακόμα. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στον ορίζοντα 2020. Γι' αυτό υποστηρίζω τα προγράμματα για τις μικρομεσαίες όπως είναι το COSME αύξηση 2,3%. Καλά δεν είναι και κανένα τεράστιο ποσοστό αυτό, ε, δεδομένων και των απορρίψεων που έχουμε. Αλλά πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, υποβάλλουν αιτήσει με καλά έργα. Όταν είναι καλά τα έργα και οι προτάσεις, είναι αυτό πολύ σημαντικό για ε, την ανταγωνιστικότητα. Και για να επανέλθω λίγο στη μετανάστευση και την ασφάλεια, είναι από τις προτεραιότητες που έχουμε αυτό το καιρό και μάλιστα πολύ ψηλά. Και οι διάφοροι οργανισμοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα χρειάζονται υποστήριξη. Γι' αυτό χαίρομαι που το EU LISA έχει περισσότερη ε, πρικοδότηση, γιατί είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να ανταποκριθεί με το προσωπικό που έχει στο έργο της. Επίσης ε, με εκπλήσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται με το Eurojust. Τους αφαιρούν έξι θέσεις υπαλλήλων. Και πώς θα δοθεί η δικαστική ε, συνέχεια όταν αφαιρείς έξι υπαλλήλους από τη Eurojust, πώς θα διεκπαιρώνουν στη Europol που έχει και όλη την τρομοκρατία και ε, όλη την ε, ανταλλαγή πληροφοριών και εκεί έχουμε βάλει πέντε θέσεις υπαλλήλων. Και έχουμε και άλλους δύο οργανισμούς όπου χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή το ΑΜΙΦ έχετε δίκιο, το Ταμείο για τη Μετανάστευση. Ελπίζω να βρεθεί κάποια συμφωνία και να ορθοποδήσει αυτή η προσπάθεια. Γιατί η ώρα δεν είναι 12 παρα 5, είναι 12 και 5. Και θα χρειαστούμε αυτή και τα 460 εκατομμύρια για το Δουβλίνο, αλλά και τα 170 ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Τώρα, οι άλλες προτάσει κομισιών, το πρόγραμμα Interrail, για να έχουν οι νέοι τη δυνατότητα να γνωρίζουν την Ευρώπη και θα συνεχιστεί το 2019 και το 2020 και κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον. Ε, μια κοινοπραξία για ε, ηλεκτρονικούς ε, υπολογιστές υψηλού επίπεδου για την ε, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ συνάδελφε Βιώτη θα τα ξαναπούμε, έχουμε να συγκρουστούμε και με τα κράτη-μέλη αρκετά για να καταλήξουμε σε ένα λογικό προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν εμφανίζουν μεγάλη προθυμία ε, συμβιβασμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη. Καλό θα ήταν. Είναι το τελευταίος προπολογισμό ε, που θα πρέπει να τελειοποιήσει και να ψηφίσει η τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Ο κύριος Κόλμελ έχει το λόγο, αλλά δεν εδώ. Βλέπω. Ο κύριος Δεπχέ, λοιπόν. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε ο, από το στόμα σας και του Θεού ε, ταυτή όσον αφορά, ε, να πηγαίνουν, ε, όσον αφορά το να πηγαίνουν ε, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου πρέπει. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι εκτιμώ σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά του συναδέλφου Βιώτη. Νομίζω ότι οι περισσότεροι προσανατολισμοί που προτείνει είναι ε, νομίζω προσανατολισμοί που μπορούν να μας βρουν σύμφωνους ακόμη και αν σε, για ορισμένα θέματα. Θα προτιμήσαμε μία έτσι, μεγέθυνση των ποσών. Ε, εξού και οι ερωτήσεις που ε, θα θέσω. Καταρχά, το πρόγραμμα COSME, είπατε ότι είναι προτεραιότητα, είναι προτεραιότητα για την ομάδα μου, ε, την ομάδα των φιλελευθέρων, οπότε θα θέλαμε μία περισσότερη προσπάθεια να γίνει. Δεν μπορούμε να δεχθούμε, εν πάση περιπτώσει, τη μείωση όσον αφορά ε, τις πιστώσει πληρωμών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Erasmus Plus. είναι προτεραιότητα και πρέπει να διευρυνθεί και για, στου, και για τους μαθητευόμενους. Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά θα, θα καταθέσουμε και σχετικές ε, ε, τροπολογίες όσον αφορά ε, τώρα κάποια ζητήματα αρχών ε, που δεν σέβεται πάντοτε η Επιτροπή μας. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να γίνεται με νέους πόρους η χρηματοδότηση των νέων προγραμμάτων και όχι με νέου ανάπτυξη άλλων ποσών. Ε, όσον αφορά το πρόγραμμα ανάπτυξης, ε, βιομηχανικής ανάπτυξης στο τομέα της άμυνας, είπαμε ότι θα γίνει μια ε, νέα χρήση ποσών, μια νέα ανάθεση ποσών ήδη υπαρχόντων. Τρεις ακόμη παρατηρήσεις για ανακατανομή των ποσών. Ε, Τρει ακόμη παρατηρήσεις. Όσον αφορά την ε, απασχόληση των νέων, ε, υπάρχει μία μείωση 33,3% σε σχέση με το 2018, σε σχέση με την τη διευκόλυνση για την απασχόληση των νέων. Νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε αυτό για να δούμε ποιο είναι το επίπεδο στο οποίο πρέπει να ορίσουμε τις απαιτήσει μας. Έχουμε ένα πιο σοβαρό πρόβλημα όμως που αφορά την κατηγορία 2 διαπιστώνουμε ότι για τον προπολογισμό του 2019, η πρόταση που γίνεται για τον προπολογισμό του 2019, οι πιστώσεις που αφορούν την προστασία του κλίματος θα είναι η 20,1% του προπολογισμού δηλαδή 0,1% πάνω από το στόχο. Αν όμως κάνουμε τον υπολογισμό για το σύνολο της περίοδου 2014 έως 2020, βλέπουμε ότι για το σύνολο της περίοδου δεν θα ισχύει αυτό δεν, δεν ισχύει αυτή η αύξηση. Δηλαδή 20% για το 2019, αλλά δεν σεβόμαστε το στόχο να έχουμε πετύχει το 20% σε όλο το πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου από το 2014 στο 2020. Το ζήτημα δεν είναι υποχρεωτικά να ενισχύσουμε κάποιες γραμμές προπολογισμού ώστε να μπορούμε να ε, πλησιάσουμε το γενικό στόχο του 20% ε, των πιστώσεων που πρέπει να αφιερώνονται ε, στην αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής και του κλίματος ε, και της θέρμανσης του πλανήτη, συγγνώμη. πράγματι καλό είναι να υπάρχει μια επισκόπηση των αναγκών. Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες για για τον οποίο η ενίσχυση είναι απαραίτητη και πάρα πολύ ε, σημαντική. Η μία είναι η Frontex, γιατί το ζήτημα του ελέγχου των συνόρων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα με τεράστιους κίνδυνους απασταθεροποίησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η ΕΑΖΟ για την δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρωπόλ και της Ευρωπόλ για την ενίσχυση της ε, συνεργασίας αστυνομικής και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Μία τελευταία ερώτηση έχω να θέσω σε σχέση με την κατηγορία 3 και επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Προτείνουμε μία επιπλέον ε, ενίσχυση της Ελλάδας 175 ε, εκατομμύρια. Τίποτε για την Ιταλία ή δεν το διάβασα καλά. Δεν, δεν, δεν ζητήσαμε τίποτα. Α, εσύ είσαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έλεγξες. Α, το έλεγξες. Μάλιστα. Καλά, θα την ε, επαληθεύσω την, την απάντησή σου. Όσον αφορά την κατηγορία 4 τώρα, ένα σύντομο σχόλιο. Ζητήσαμε από όλα τα όργανα να κάνουν ε, μία μείωση 5% του προσωπικού τους εδώ και πολλά χρόνια. Ε, διάβασα μία έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και λέει ότι, πολύ εκπληκτικό είναι αυτό, ότι κατά τη διάρκεια αυτή, της, αυτή, της περίοδου αυτή, ο αριθμός των προσωρινά απασχολούμενων ή με άλλο καθεστώς έχει αυξηθεί, ότι φυσικά έχει αυξηθεί ε, το ποσό των ε, μισθών κατά 9% αν θυμάμαι καλά. Ε, δεν θα ήθελα να ξαναπάμε προς τα πίσω και να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά πραγματικά προβληματίζομαι κατά πόσο έχει έχει νόημα αυτό που αποφασίσαμε. Κάτι ακόμη που αφορά την Τουρκία. Ε, η ομάδα μου πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να χρηματοδοτήσουμε αφορά, ό,τι αφορά τη διευκόλυνση για την Τουρκία. Είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα όχι μόνο των μεταναστευτικών ροών αλλά και της πολιτικής ε, κατάστασης ε, της Ευρώπης, ειδικότερα όσον αφορά τώρα τα ποσά τις πιστώσεις που αφορούν την ένταξη της Τουρκίας έχω πραγματικά σοβαρά ερωτηματικά να εκφράσω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για τις παρατηρήσεις αυτές. Η κυρία Νιριάντα δεν είναι παρούσα, ο σκιώδης της Γκουε, ο κύριος Τάραντ επίσης. ούτε ο εκπρόσωπος FDD είναι εδώ, αλλά ο κύριος Κόλμπελ ε, ξαναμπήκε στην αίθουσα, ίσως θα μπορούσε να μας παρουσιάσει και αυτό τις σκέψεις του για την έκθεση ε, διότι για την εντολή στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου της 12ης Ιουλίου, της προπαρασκευαστικής φάσης δηλαδή, της διαβούλευσης για τον προϋπολογισμό του 19. Όχι, δεν έχει να πει κάτι. Οπότε παίρνει το λόγο ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Βιώτη. Καλά έχετε επιλέξει το κέντρο βάρους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο όταν λειτουργούν οι επιχειρήσεις και υπάρχει αρκετή δουλειά, ε, τότε έχουμε και φορολογικά έσοδα και μπορούν να υποστηριχθούν όλα αυτά τα προγράμματα ε, που είναι όλο και πιο σημαντικότερα για το μέλλον. Και η συνάδελφος Χολμάιερ μίλησε για τη Eurojust που είναι τεράστιο θέμα ε, που θα βρούμε μπροστά μας και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Βλέπουμε και ότι η συνεργασία δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά ή όπως θα θέλαμε, στην ενίσα και στην προστασία των δεδομένων. Καλό θα ήταν να το ε, ενώσουμε με την ΕΣΑ και με τον ΠΕΡΕΚ. Αυτή η οριζόντια επικοινωνία είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα ε, έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Επίσης, υπάρχει η ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη που θα πρέπει να πιάνει τόπο για τους Ευρωπαίους πολίτες και να παρέχει προστιθέμενη αξία. Αυτή η διευκόλυνση λοιπόν, ΣΕΦ, βεβαίως είναι και ένα επενδυτικό πρόγραμμα για δημιουργία θέσεων εργασίας και όλα αυτά τα προγράμματα αποδίδουν και ε, οτιδήποτε έχει να κάνει με παραγωγή πλούτου παράγει και έσοδα φορολογικά που μπορεί στη συνέχεια να δώσει κανείς για την ε, άμυνα και λοιπά και το, το σώμα αλληλεγγύης και όλα αυτά που είναι σημαντικά για το μέλλον. Ένα τελευταίο που θέλω να αναφέρω και ενδιαφέρει και το ΕΛΚ, το Horizon 2020. Για μας είναι πολύ σημαντικό στο πρόγραμμα αυτό να ε, εκπέμψουμε κάποια μηνύματα ότι η Ευρώπη στο διεθνή ανταγωνισμό είναι παρούσα και δεν ε, εγκαταλείπει. Είδαμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας με νομπελίστες ε, πραγματικά έχουμε καλύψει το κενό που είχαμε ή την απόσταση και μπορούμε να δείξουμε ότι και το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται να αποτελέσει αυτό ένα κέντρο βάρους μαζί με το Erasmus Plus. Ε, είναι αυτά τα προγράμματα που ε, ενδιαφέρουν περισσότερο τους νέους και τους κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Όπως και το πρόγραμμα Wi-Fi for You Ακριβώς υποστηρίζουμε τον εισηγητή και είναι πολύ σημαντικό τώρα να βγούμε, να υπερασπιστούμε όλα αυτά και να τα διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Και με συνέπεια. Ευχαριστώ κύριε Ρίμπιχ. Οπότε, εδώ είμαστε στο τρίτο τμήμα, όχι στα υπόλοιπα τμήματα. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Όχι. Δεν βλέπω. Προσωπικά, πιστεύω ότι η Οδύσσια του πλοίου Ακουάριος θα κάνει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν ορισμένες προτεραιότητες στον προϋπολογισμό για το 2019. Για την απασχόληση των νέων, θα ρωτήσω, μάλλον το γενικό μας εισηγητή, αν μπορούμε να ε, διοχετεύσουμε τις πιστώσεις σε πιο διαρθρωτικά μέτρα, δηλαδή επαγγελματική κατάρτιση και μαθητεία. Γιατί αυτά είναι εκείνα που επιτρέπουν να, καταπολεμούμε αποτελεσματικά την αναργία των νέων, γιατί είναι διαρθρωτικά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις πιστώσεις στοχευμένα. Και βλέπω και το Ταμείο για την Ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας είχε κάποιες επενδύσεις και μήπως είναι ευκαιρία αυτή να υπογραμμίσουμε ότι Εάν δαπανούμε κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για την Άμυνα, θα μπορούσαμε να κάνουμε οικονομίες στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αν δηλαδή γίνει πιο ουσιαστικός ο ευρωπαϊκός αμυντικός προϋπολογισμός, θα μπορούσαμε να έχουμε λιγότερες αμυντικές δαπάνες από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την ενδεχόμενη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Νομίζω είναι ένα αρκετά καλό επιχείρημα για να ενισχύσουμε αυτή την επιθυμία για το, τον πόθο για την Ευρώπη και να αποκτήσει και πάλι την έγκλη της Ευρώπης. Μήπως θα μπορούσε να μας πει τώρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψή της, ο κύριος Ρέλ. Τι έχετε να πείτε για την Οδύσσια του Ακουάριος. Ο κύριος Ρέλ έχετε αναθεωρήσει κάπως τα κονδύλια του προπολογισμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Clear. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι όποιος παρακολουθεί τη συζήτηση αυτή να δει ότι το θέμα της αλληλεγγύης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα της μετανάστευσης είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση σοβαρή η οποία μέχρι τώρα δεν έχει οδηγήσει σε κάποια συνένεση στο Συμβούλιο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο 2. Συνεπώς λοιπόν το Συμβούλιο θα πρέπει να παρακολουθήσει προσεκτικά την εξέλιξη της συζήτησης και αν είναι απαραίτητο να αναθεωρήσει κάποιες προτάσεις ή να κάνει μια ανακατανομή δημοσιονομικών μέσων. Δεν φτάσαμε στην φάση αυτή, αλλά παρακολουθούμε καλά τις συζητήσεις προσεκτικά. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια επικοδομητική στάση στα πλαίσια της έκθεσης της σύνταξης, της σύνταξης της έκθεσης του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε τεχνικό επίπεδο ε, στη διάθεσή του. Να τελειώσω εδώ με κάποιες επιμέρους πρακτικές λεπτομέρειες τις οποίες έχουμε προσπαθήσει εμείς να ενσταλάξουμε στην ε, έκθεση, στην πρόταση έκθεσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροπολόγηση του κοινωνικού κανονισμού για την πρωτοβουλία για τους νέους υπάρχει μια χρονική προθεσμία για την αποδοχή της πρότασης αυτής από την Επιτροπή είναι η 26η Ιουνίου. Σχετικά τώρα με την συνεχιζόμενη αξιολόγηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των σημαντικών ποσών των πιθανών πιλωτικών και προπαρασκευαστικών προγραμμάτων και δράσεων που έχουν υποβληθεί από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για προκαταρκτική ανάλυση, όπως φαντάζεστε, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει αρχίσει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είμαστε ικανοί να δώσουμε την προκαταρκτική μας αξιολόγηση στο τέλος του μήνος Ιουνίου. πριν δηλαδή από τον διάλογο της 12ης Ιουλίου και μια τελευταία πληροφορία τώρα που η πολιτική συμφωνία έχει πλέον επιτευχθεί και στον τομέα της πρωτοβουλίας για την άμυνα και σε σχέση με το σώμα αλληλεγγύους. Οι δημοσιονομικές συνέπειες αυτών των δύο συμφωνιών θα πρέπει να ενσωματωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια διορθωτική επιστολή η οποία θα ακολουθήσει δυστυχώς την συνάντηση της 12ης Ιουλίου. Ευχαριστώ κύριε Ουρέλ για να κλείσουμε. Κύριε Βιώτη, έχετε ξανά το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά θερμά τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για τα σχόλιά τους που είναι πολύ χρήσιμα για μένα. αν πρέπει να κάνω μία αξιολόγηση πολιτικού τύπου και λιγότερο τεχνικού τύπου από αυτά τα οποία είπα στην εισαγωγή, έχω την αίσθηση ότι οι τροπολογίες τις οποίες θα καταθέσουν οι πολιτικές ομάδες η προθεσμία είναι αύριο μεθαύριο και θα προσπαθήσουμε την επόμενη εβδομάδα να βρούμε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις, κάτι το οποίο θα προσπαθήσει με τη σειρά του να καταστήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρη με συγκεκριμένους στόχους. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει με το Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και με το Συμβούλιο αυτά τα οποία ακούσαμε και για τη μετανάστευση και αυτά τα οποία είπε και η κυρία Χολμάιερ ε, για την υπόθεση του Ακοάριους ε, είναι παράλογο να περιμένει κανείς να υπάρξει ένα επεισόδιο ευτυχώς αυτή τη φορά όχι τραγικό για να αφυπνιστεί η συνείδηση των λαών μας, των χωρών μας αλλά αν αυτό κάτι μας μάθει είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει και το Συμβούλιο να κατανοήσει ότι αν θέλουν να δίδουν αυτή τη βοήθεια, αν θέλουν να υπάρχουν λιγότερες αναχωρήσεις και λιγότερα σκάφη, θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην Αφρική. Και για να επενδύσουν περισσότερο στην Αφρική απαιτούνται περισσότερα χρήματα στον προϋπολογισμό. Ε, αυτό αυτό λοιπόν είναι που θα βοηθήσει τους πολίτες, αυτό που θα βοηθήσει τους κυβερνώντες, δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει και αυτή τις δικές της προτάσεις, έτσι ώστε κάποια χρήματα να μην επενδύονται στην Ευρώπη, αλλά να επενδυθούν αν είναι δυνατόν στην Αφρική. Ελπίζω να καταλήξουμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια λογική πρόταση συνολικά. Εγώ δεν αναφέρθηκα στα της Ιταλίας και λόγω της σύγκρουσης αν θέλετε των ιδιωτήτων τις οποίες έχω αλλά οι συνάδελφοι από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα ε, δεν έχω πάρει ακόμα τις προτάσεις τους για να μπορέσω να τις σχολιάσω. Τώρα για τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία τέθηκαν για το Interrail, για το Horizon 2020 κτλ. Νομίζω ότι εγώ θα πρέπει να περιμένω τις τροπολογίες σας και θα προσπαθήσουμε να τις ενσημετώσουμε. Θα ήθελα και εγώ όπως ο κύριος Ρομπίχ να θεωρήσω ότι ε, ο τελευταίος προϋπολογισμός αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου να είναι ένας προϋπολογισμός για τους νέους, για τα συμφέροντα των νέων, για το μέλλον των νέων. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια συζήτηση στην Επιτροπή μας, στο Κοινοβούλιο γενικά, στη συνεργασία και τον διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και επίσης θα πρέπει και εμείς με τις κυβερνήσεις μας στις χώρες μας να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους διερμηνείς οι οποίοι βρίσκονται σε μια κάποια αναταραχή τις τελευταίες εβδομάδες. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγητά για αυτά τα ελπιδοφόρα λόγια σας που θα μαγέψουν και πάλι την Ευρώπη. Λοιπόν, τούτων όλων λεχθέντων. Τροπολογίες για τη σχέδια έκθεση του κυρίου Βιώτη μπορείτε να κάνετε μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, απόψε. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 28 Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή. λήξη της συνεδρίασης πριν τις 12.30. Ευχαριστούμε του διερμηνείς για τη συμμετοχή του. Ελπίζουμε να καταλήξουν κάπου συνομιλίε. Αν δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο, διακόπτει τη συνεδρίαση. Reprise à 14h30. Συνέχεια στις 2.30.